Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, τα πρακτικά της Συνόδου της 8ης Ιουλίου για τα οποία σας ρωτώ αν έχετε κάποια παρατήρηση ή ένσταση. Από ό,τι βλέπω, όχι επομένω ε, εγκρίνονται. Η